Oh, Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη και αρχίζουμε σχεδόν στην ώρα μας. Είναι η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο. Και καλωσορίζω τον Υπουργό στον παρθενικό του γύρο ερωτήσεων με την Ισπανική Προεδρία. Θα πάρουμε τα ερωτήματα με τη σειρά που εμφανίζονται. Η πρώτη ερώτηση του κυρίου Ατόντο κρίθηκε μη παραδεκτή γιατί αφορούσε το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο ένα θέμα που συζητήθηκε χθε την Τρίτη. Οπότε περνούμε στην δεύτερη ερώτηση του κυρίου Γκάι Μίτσελ με θέμα τη μείωση της προσφοράς πιστώσεων και δανείων για τις επιχειρήσεις. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. η εξασφάλιση της επαρκούς πρόσβασης των επιχειρήσεων στη δανειοδότηση και οι σχετικές δράσεις των κρατών μελών είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ και καιρό το Συμβούλιο και το γνωρίζετε. Πέρυσι τον Ιανουάριο το Συμβούλιο παρατήρησε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν πιο αποφασιστικές δράσεις για να απεμπλέξουν μεταξύ άλλων τις ε, αγορές του δανεισμού και των πιστώσεων. Και την Άνοιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διακήρυξε την ανάγκη συνέχισης των μέτρων οικονομικής ανάκαμψης και κάλεσε την ε, Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των ελλημένων αποφάσεων και να ενημερώσουν σχετικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου έγινε η αξιολόγηση των ε, μέτρων που ενέκριναν τα κράτη-μέλη για την υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού κλάδου και τη συμβολή του στη σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής περιλήφθηκαν σε μια έκθεση που υπευλήθη ε, από το Συμβούλιο Υπουργών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην έκθεση αυτή το μήνυμα ήταν θετικό. Επισημάνθηκε δηλαδή ότι υπήρξαν εχέγγυα και μηχανισμοί κεφαλαιοποίησης στα κράτη-μέλη χάρη στα μέτρα που εγκρίθηκαν και ήταν σημαντική η συμβολή των κρατομένων προκειμένου να αντιστραφεί αυτός ο φαύλος κύκλος. Γιατί στα τέλη του 2008 υπήρξε κίνδυνος ε, κατάρρευσης ε, του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Υπήρξαν λοιπόν θετικές συνέπειες ε, για την βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και στο δανεισμό. Το Συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι τα ελιμένα από τα κράτη μέτρα ήταν σημαντικά για να ξανανοίξουν η κρουνοί του δανεισμού. Βέβαια, ο τραπεζικός κλάδος υφίσταται αρκετές πιέσεις για το θέμα αυτό. Γι' αυτό και το Συμβούλιο τότε ζήτησε από τα κράτη-μέλη να προβούν σε κατάλληλες κεφαλαιοποίησεις ή στην εξασφάλιση ισορροπίας για να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση των επιχειρήσεων στο δανεισμό. Και πέρυσι το Δεκέμβριο το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι τα κράτη-μέλη είχαν εφαρμόσει ε, μια ευρύτατη δέσμη μέτρων υποστήριξης για να εξασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και διαπίστωσε παρόλα αυτά ότι η ανάκαμψη δεν ήταν ακόμη η αναμενόμενη. Γι' αυτό και θα πρέπει στρατηγικά να προβλεφθούν νέα κεφάλαια και σταδιακά για να συνεχιστεί η δυνατότητα πρόσβαση στο δανεισμό. Οπότε και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρακολούθησαν την εφαρμογή αυτών των μέτρων και δόθηκαν κάποιοι προσανατολισμοί με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η κατάσταση χάρη και στη συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και έτσι η, η πρόσβαση στο δανεισμό για τις επιχειρήσεις έγινε καλύτερη και η τραπεζική ρευστότητα επίσης βελτιώθηκε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Είμαι βέβαιος ότι... Είμαι βεβαίω ότι ο κύριος Γκάι Μίτσελ θα έχει και συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Υπουργό για την απάντησή του. Να πω στον Υπουργό ότι με βάση την εμπειρία μου ορισμένες τράπεζες, όχι όλες βεβαίω, αλλά ορισμένες, ίσως και πολλές, ε, συμπεριφέρθηκαν ανεύθυνα κατά τη διάρκεια ε, ε της, της ανάπτυξης αγορά αγοράς και ορισμένες τράπεζε, πολλές τράπεζε, μάλιστα, εξακολουθούν να συμπεριφέρονται ανεύθυνα. και, και κατά την κρίση αλλά και κατά την περίοδο της ανάκαψης. Για παράδειγμα, στο Δουβλίνο, μία συγκεκριμένη εταιρεία ε, ε, η οποία ε, είχε πολύ υγιή διαχείριση και εκπλήρωνε τις, τις, τις, τις, τις υποχρεώσεις του απόλυτα ο διαχειριστής και όμως το περιόρισαν τη δυνατότητα υπερανάληψης. Δεν έπρεπε λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο. Σας παρακαλούμε πείτε στις τράπεζες ότι χρησιμοποιούν τα χρήματα των φορολογμένων και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο συμφέρον και όχι μόνο το συμφέρον των μετόχων τους. Γιατί ορισμένοι από τους μετόχους αυτούς είναι και ιδιαίτερα πλούσιοι. Ευχαριστώ. Να σα υπενθυμίσω σε όλου ότι ε, η συμπληρωματική ερώτηση είναι ε, για μισό λεπτό και, ε, και όχι παραπάνω. Υπουργέ, αν θέλετε να απαντήσετε. Ναι, ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για τη συμπληρωματική ερώτηση. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι από την άποψη του Συμβουλίου και των Ευρωπαϊκών Θεσμών νομίζω ότι υπήρξε σωστή δράση ε, και υπήρξε ε, δράση έτσι ώστε να μην καταρρεύσει η οικονομία. Το ε, Συμβούλιο Εκοφήν παρακολουθεί και εξακολούθησε να παρακολουθεί τα μέτρα που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη, το κάνει αυτό σε συστηματική βάση. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή το Εκοφήν εξετάζει με ποιο τρόπο, με ποιο, με, πώς μάλλον χρησιμοποιούνται αυτές οι εγγυήσεις, κατά πόσον υπάρχουν περιορισμοί σε ορισμένες επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και πώς ε, ολοκληρώνεται η χρηματοδότηση εκ μέρους ε, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ε, ότι στις 7 Δεκεμβρίου 2009 ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Τρισέ, είπε ότι, ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς την προσφορά. Δηλαδή δεν υπάρχουν περιορισμοί στην προσφορά. Αν υπάρχουν τράπεζες ε, ε, που ακολουθούν άλλη τακτική, τότε αυτό έχει να κάνει με το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Αλλά εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν υπάρχει κανένα είδος περιορισμού. Πάντως, ε, είναι φυσικό ότι το Συμβούλιο μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να εξετάσει ε, και υπάρχουν και οι κατάλληλε οδηγίε ε, που θα ζητηθούν στα πλαίσια τη χρηματοπιστωτική εποπτεία και θα εξετάσουμε και οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία που τυχόν προτείνει η Επιτροπή προ την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστούμε. Σα ευχαριστώ. Δεν έχω άλλη συμπληρωματική ερώτηση. Συμπληρωματική ερώτηση για αυτό το θέμα. Ναι, κυρία Κρίς, κοιτάξτε, μία από τις προτεραιότητες ε, της ε, Προεδρίας Συμβουλίου είναι η ενίσχυση της επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή και κυρίως στη Λατινική Αμερική. Αλλά για ποια επιρροή μιλάμε. Ε, ε Όπω έχουν τα πράγματα σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Συμβούλιο θα ήθελε μέσω των συμφωνιών ελεύθερη συναλλαγή ε, να εξετάσει τι γίνεται με τα καθεστώτα τα οποία, ε, ε, όπου υπάρχει πρόβλημα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για παράδειγμα, το, το, οι εξελίξει και τα γεγονότα στο Περού. Εκεί βλέπουμε σαφώ πώ συνεργάζεται η κυβέρνηση με τι πολυεθνικέ και το πώ προβαίνει σε δίμευση των περιουσιών των αυτοχθόνων. Άλλο παράδειγμα, το παράδειγμα τη Κολομβίας. Μια χώρα ε, όπου δολοφονούνται διαρκώς οι συνδικαλιστές. Ρωτώ λοιπόν, τι θα γίνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και πώς ε, εντάσσεται στο πλαίσιο τη εξωτερική πολιτική προς τη Λατινική Αμερική. Σας ζητώ συγγνώμη, λέει η κυρία Γουόλης, αλλά τι σχέση έχει η ερώτησή σας με την τελευταία αυτή ερώτηση που έγινε. Δεν ξέρω αν έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν στην ώρα των ερωτήσεων. Η συμπληρωματική ερώτηση πάντω έχει να κάνει με τη βασική ερώτηση. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε την ερώτησή σα. Είναι εκτό διαδικασία. Σα προτείνω, αν έχετε την καλοσύνη, να κοιτάξετε του κανόνε. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, δεν υπάρχουν συμπληρωματικέ ερωτήσει. Έκλεισε λοιπόν ε, η συζήτηση για την προηγούμενη ερώτηση. Θα συνεχίσω λοιπόν. Εκτός και αν υπάρχει άλλη ερώτηση συμπληρωματική αναφορικά με το θέμα των ε, πιστώσεων και των δανείων για τις επιχειρήσεις. Κυρία και και για πείτε μας. 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας. Ναι, περί αυτού πρόκειται. Έχω και εγώ συμπληρωματική ερώτηση για το ίδιο θέμα. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική στα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τη βοήθεια στις επιχειρήσεις, θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση για την κατάσταση στην Ελλάδα. Γιατί εκεί είναι που αντιμετωπίζεται μία δίνη κρίση. Εκεί, στην Ελλάδα, προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις, ειδικέ δράσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Νομίζω ότι για το ίδιο θέμα υπάρχει η επόμενη ερώτηση Οπότε θα παρακαλούσα τον Ευρωβουλευτή να περιμένει όταν φτάσουμε εκείνη, σε εκείνη την ερώτηση, γιατί εκεί θα δώσω απάντηση για την Ελλάδα. Γιατί ακριβώς υπάρχει συγκεκριμένη ερώτηση για την κατάσταση στην Ελλάδα. Περιμένετε λοιπόν λίγο αργότερα. Can you say to which question... σε, σε ποια ερώτηση αναφέρεστε κύριε Υπουργέ, ώστε να ξέρει ο Ευρωβουλευτής μέχρι πότε θα πρέπει να περιμένει για την απάντηση είναι η ερώτηση 9 στον κατάλογο που έχω εγώ. Η 8, μια και η πρώτη αφαιρέθηκε. Είναι η ερώτηση της κυρίας Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου που αφορά την δημοσιονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Μάλιστα λοιπόν, επειδή και ο βουλευτής που έθεσε την ερώτηση αποδέχεται την απάντηση σε μετέπειτα χρονικό σημείο, να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. του κυρίου Πόσελτ για την ε, προσχώρηση του Κωσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπουργέ, όποτε θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο επανέλαβε τους προσανατολισμούς εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής γειτονίας αλλά και της πολιτικής διεύρυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν ανέκαθεν της γνώμης ότι τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν μια ευρωπαϊκή προοπτική και μια ενταξιακή προοπτική. Και μάλιστα στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2009 επιβεβαιώθηκε η ανάγκη εκπλήρωσης κάποιων ισότιμων προϋποθέσεων για την διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης των Δυτικών Βαλκανίων. Σε ό,τι αφορά το Κωσυφοπαίδιο συγκεκριμένα, το Συμβούλιο παρατηρήσε ότι στην περίπτωση αυτή τα κράτη-μέλη αποφάζαν με βάση την εθνική τους πρακτική και το διεθνές δίκαιο. Και μάλιστα η μονομερής διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κωσυφοπεδίου αποτελεί το αντικείμενο προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο. Πάντως το Συμβούλιο δεν αγνόησε το Κωσυφοπέδιο στην πολιτική για τα Βαλκάνια και υπήρξε συνένεση μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών μελών για το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Υπάρχει τέτοια διευκόλυνση και για το κοσυφοπαίδιο. Και μάλιστα έγινε δεκτή με ικανοποίηση ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέματα μέσα ενίσχυσης ε, της ε, πολιτικής και κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης του κοσυφοπαιδίου. Το Συμβούλιο προσκάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την παρότερη να λάβει τα μέτρα για να στηρίξει την προσέγγιση του κοσυφοπεδίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιώντας ε, αυτή την ε, ευρωπαϊκή προοπτική. Και μάλιστα το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμπλέξει και το κωσυφοπέδιο στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στα και στην ε, ενεργοποίηση του μηχανισμού για το πρωταξιακό μέτρο και στις διαπραγματεύσεις για, τον, για τη Συμφωνία Σύνδεσης. Και μάλιστα όλα αυτά τα συμπεράσματα συμπεριλήφθηκαν και στο τελευταίο Συμβούλιο της 10 ε, και 10 η Δεκεμβρίου του 2009. Ευχαριστώ κύριε Σπόσελτ, ευχαριστώ Υπουργέ. Δύο συγκεκριμένα στοιχεία ήθελα να θέσω. Καταρχάς, πιστεύετε ότι υπό την Ισπανική Προεδρία θα πετύχουμε κάτι να κινήσουμε κάτι σε ό,τι αφορά το καθεστώ των θεωρήσεων για να μην παραμείνει σε φυλακή στα ελεύθερα Βαλκάνια το Κωσυφοπαίδιο και κατά δεύτερον τι θα κάνετε με τα κράτη-μέλη που δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα το κοσυφοπέδιο προκειμένου να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή αλλά καταρχάς σε ό,τι αφορά το καθεστώς θεωρήσεων ο υπουργό, λέει η Πρόεδρος. Ναι, αναφέρθηκε στη διευκόλυνση των θεωρήσεων προηγουμένως. Το Συμβούλιο ήταν ανέκαθεν της γνώμης ότι και το 25 θα πρέπει να επωφεληθεί από το καθεστώς των θεωρήσεων αν υπήρχε απελευθέρωση για όλη την περιοχή. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με τις λεπτομέρειες αυτής της πρότασης. Πρώτα θα γίνει μια διευκόλυνση των θεωρήσεων και κατόπιν μια απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης και πρώτα θα επεξεργαστεί αυτές τις προτάσεις και μετά θα υποβάλει σχετική πρόταση στο Συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις ενδιαφερόμενες χώρες, ε, εμπροκειμένο με το κοσυφοπαίδιο και ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο. Τώρα η ιδέα της ε, κατάργησης των θεωρήσεων που διευρύνεται στις γειτονικέ χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια ιδέα που βρίσκει σύμφωνα το Συμβούλιο και την Ισπανική Προεδρία και είναι και ένας από τους βασικούς πολιτικούς προσανατολισμούς που θα προωθήσουμε στο εξάμεινό μας στην Ευρώπη. Δηλαδή θέλουμε να διευκολύνουμε την κινητικότητα και την ε, δυνατότητα κυκλοφορίας, διακίνησης και επικοινωνίας όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μεταξύ των γειτονικών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί νομίζω ότι είναι αμοιβαίως επωφελής μια τέτοια τακτική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που απαλλάσσει από την υποχρέωση ε, θεωρήσεων, αλλά και τις χώρες αυτές που φυσικά ε, εφαρμόζουν καθεστώς αμοιβαιότητας. Η ε, επερωτήσει μπορώ να επιτρέψω και έλαβα πολλές αιτήσει από την κυρία Μότσα και από τον κύριο Χουντή. Και θα ακούσουμε και τις δύο ερωτήσει και μετά θα απαντήσει ο Υπουργός, η κυρία, ο κύριος Μόλτσο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Με όλες τις πρωτοβουλίες που προγραμματίζει το Συμβούλιο για το Κωσυφοπέδιο θα ληφθεί υπόψη και η Σερβία, γιατί η Σερβία είναι ένα κεντρικό κράτος για την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε όλα τα βήματα. Ευχαριστώ, κύριε Χουντής. Κύριε Υπουργέ, εκτιμώ θετικά τη στάση της χώρας σας, της Ισπανίας, που δεν έχει προχωρήσει στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Κωσυφοπεδίου και την πρόσφατη απόφασή σα να αποσυρθούν τα ισπανικά στρατεύματα που στράτευαν μέχρι τώρα στο κωσυφοπαίδιο. επειδή είμαστε και σε περίοδο οικονομικής κρίσης θα σας κάνω την πεζή ερώτηση πόσο κόστιζαν στην ισπανία αν είσαστε εύκολο να μου δώσετε το στοιχείο πόσο κόστιζαν η παραμονή αυτών των στρατευμάτων και αν μπορείτε να σχολιάσετε τη στάση τη δική μου χώρα της ελλάδας που έχει την ίδια δύναμη στο κωσυφοπαίδιο με γνωστά τα οικονομικά προβλήματα αν είναι σωστό να παραμένουν εκεί τα στρατεύματα στο κωσυφοπαίδιο. ευχαριστώ πολύ. σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση για τη σερβία φυσικά η Σερβία σίγουρα είναι η ισχυρότερη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων και θα πρέπει να την λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε πολιτική και σε οποιαδήποτε ενταξιακή προοπτική. Γιατί αυτή είναι η ευρωπαϊκή πολιτική για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και υπάρχει μια πρόσφατη συμφωνία, θα τη γνωρίζετε, για την απελευθέρωση των θεωρήσεων σε ό,τι αφορά τη Σερβία. Μια κατάργηση των θεωρήσεων. Και πολύ πρόσφατα, μετά τη, την απελευθέρωση των διαπραγματεύσεων για την ενδιάμεση συμφωνία της Σερβίας υπήρξε και η επίσημη αίτηση υποψηφιότητας της Σερβίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ε, είμαστε υπέρ της ε, νομοθεσίας, υπέρ της εφαρμογής της νομοθεσία, ε, θα επιληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εξετάσει την κατάσταση και θα προτείνει την πιθανότητα ένταξη τη Σερβία και την ένταξη μια ενταξιακή διαδικασία εφόσον πληρούνται τα κριτήρια τη Κοπεχάγη. Γιατί σίγουρα η Σερβία έχει αναμφισβήτητο βάρο στα Δυτικά Βαλκάνια και κατά τη γνώμη μα και η Σερβία έχει ενταξιακή ευρωπαϊκή προοπτική. Και μάλιστα στην περίπτωση αυτή η ομοφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν υπέρ τη απεμπλοκή τη ενδιάμεση συμφωνία ε, για τι διαπραγματεύσει με την ε, Σερβία. Κύριε Ευρωβουλευτά, μου θέσετε μια ερώτηση που σχετίζεται με εσωτερικέ αποφάσει και εσωτερική πολιτική τη Ισπανική κυβέρνηση. Εδώ εκπροσωπώ το Συμβούλιο, όχι μια συγκεκριμένη χώρα, όχι την πατρίδα μου, αλλά ολόκληρο το Συμβούλιο Υπουργών. Και δεν έχω τέτοια ακριβή στοιχεία σαν αυτά που μου ζητήσατε. Είναι πολύ δύσκολο να βρω τα στοιχεία αυτά για το κόστο που ζητήσατε. Δεν νομίζω ότι ε, έχει νόημα να μιλήσω εδώ για μια συγκεκριμένη χώρα, γιατί εδώ εκπροσωπώ το Συμβούλιο της Ένωσης, που απαρτίζεται από 27 χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Και τώρα να περάσουμε στο επόμενο ερώτημα του κυρίου Higgins αναφορικά με την καταστροφή των τροπικών δασών. Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός. Ναι, ε, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι το Συμβούλιο συμφωνεί ιδιαίτερα μαζί σας, κύριε Χίγγινς. Συμφωνούμε στο ότι η γεωργία και η καταστροφή των δασών αποτελούν συγκεκριμένους παράγοντες ε, που συνδέονται άμεσα με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρωπου στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι εύκολο βέβαια να ξέρουμε ε, ποιος από τους δύο παράγοντες ε, επιβαρύνει περισσότερο τα πράγματα. Η συζήτηση αυτή βέβαια είναι περισσότερο επιστημονική φύση παρά πολιτική. Αλλά πάντω ε, να σα πω ότι θα πρέπει να δούμε και τι δύο αυτέ συνιστώσει και να δράσουμε ταυτόχρονα. Νομίζω ότι πάντα ήταν έτσι τα πράγματα. Πάντα όταν μιλούσαμε για την αηφόρο γεωργία ε, ε, εξετάζαμε και τι δύο πτυχέ. Και μάλιστα αυτό οδήγησε στην τροποποίηση τη πολιτική ε, ανάπτυξη υπαίθρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια τη μεταρρύθμιση κοινή αγροτική πολιτική. Λαμβάνεται υπόψη λοιπόν αυτό το στοιχείο για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει ε, ε, του μετριασμού και τη αντιμετώπιση κλιματική αλλαγή. Και όπω ξέρετε, στα πλαίσια τη εξέλιξη τη πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική ε, έχει κατέχει σημαντική θέση στα πλαίσια ε, της ευρύτερης πολιτικής καταπολέμησης ε, της κλιματικής αλλαγής. Ήδη από το 2008 το Συμβουλίο υποστήριξε τη θέση της Επιτροπής για την καταστροφή των δασών και επίσης να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για το ότι η μάζα των δασών που αποτελεί αντικείμενο απώλειας εάν σταματήσει μέχρι το 2030 το πολύ και μειωθεί η καταστροφή των τροπικών δασών τουλάχιστον κατά το 50% ε, σε σχέση με το 2020. Αυτή ήταν η στόχη που είχε αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό θα πρέπει να βοηθήσουμε έτσι ώστε να υπάρξει αηφόρο διαχείριση των δασών, να αντιμετωπίσουμε την αποψήλωση και την ε, υποβάθμιση των δασών. Όλα αυτά αποτελούν μέρο ε, των στόχων που έχει θέσει η Προεδρία τη Ισπανία και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ένα από τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν δηλαδή μέσα ε, για την αντιμετώπιση της καταστροφής των δασών, καθώς επίσης θα πρέπει να, εφαρμοστεί, να εφαρμοστούν οι κανόνες της διακυβέρνησης και διαχείρισης των δασών, όπου προβλέπεται η δημιουργία νομικού πλαισίου για να μην γίνεται εισαγωγή ξυλίας ε, που ε, αποτελεί αντικείμενο παράνομης υλοτομίας. Ε, αυτή είναι και η θέση μας και πρέπει να σας πω ότι ε, Βεβαίως, ε, όσον αφορά ε, τους μη εκπληρωθέντες στόχους της Κοπενχάγης και το βαθμό της απογοήτευσης που υπήρξε, ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι τονίστηκε ε, το πόσο σημαντικό είναι το θέμα της καταστροφής τροπικών δασών και το πώς αυτό πρέπει να εξεταστεί σε επίπεδο αναπτυσσόμενων χώρων σε συνδυασμό με τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Επίσης, να πούμε ότι η συνδιάσκεψη πήρε απόφαση για δράσεις για μείωση της αποψήλωσης και καταστροφής των δασών, προωθώντας ε, ε, την ε, υποστήριξη προς τις ικανότητες που έχουν οι ανεψόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριο Χίγκιν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Ισπανική πρόεδρε. Ήταν πολύ καλή η εκκίνησή σας. Βίβα Λεσπάνια λοιπόν. Να πω για την ερώτηση αυτή ότι τα δάση απορροφούν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και η τραγωδία της Βραζιλίας και επειδή ο Αμαζόνιος βρίσκεται κατά 60% στη Βραζιλία είναι η καταστροφή και τι σημαίνει αυτή δηλαδή οι τεράστιες εκτάσεις που έχουν καταστραφεί αυτό πέρα από το διοξείδιο του άνθρακα καταστρέφει πολλά είδη ζωής και από πλευρά της γεωργικής ε, παραγωγής ξέρουμε ότι τα πρότυπα γεωργικής παραγωγής δεν ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά. Τι μπορούμε να κάνουμε επί του παρόντος όμως, Πρόεδρε, μήπως απλά λόγια μπορούμε να απευθύνουμε. Το λόγο έχει ο Υπουργό. Κύριε Χίγκιν, θέλω να σα πω ότι συμφωνούμε απόλυτα με αυτά τα οποία είπατε κι εσείς. Όσον αφορά τη βιοπικιλότητα, η Ισπανική Προεδρία έχει θέσει συγκεκριμένο στόχο για την εξέταση σε βάθος ε, του θέματος ε, για την ε, αηφόρο χρήση. Δηλαδή, πρέπει να εξετάσουμε σε βάθος το θέμα της βιοποικιλότητας και που αποτελεί κεντρικό σημείο της Προεδρίας. Και σε ευχαριστώ για αυτά τα οποία είπατε και είπατε ότι ξεκινάμε καλά, ξεκινήσαμε καλά ως Προεδρία. Πάντως να σας πω ότι η Επιτροπή ε, ε, πιστεύει, μάλλον ε, μας έχει πει ότι θα παρουσιάσει στις αρχές του, του, του τρέχοντος έτους ε, μία πράσινη βίβλο για την, ένα πράσινο βιβλίο για την προστασία των δασών. Σωστό είναι αυτό. Θα εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα τα οποία πλήττουν τις περιοχές αυτές. Εσείς αναφερθήκατε σε, ορισμένα τέτοιε σε ορισμένες τέτοιες περιοχές, υπάρχουν και άλλες όμως και άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, η ζημιά που προέρχεται από τι πυρκαγιέ στα δάση. Πολλά στοιχεία λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη. Πάντω είμαι σίγουρο ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε το θέμα τη καταστροφή των δασών μα. Και βεβαίω ε, όλα αυτά στα πλαίσια και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, Το θέμα αυτό θα αποτελέσει σημαντικό σημείο, σημείο κλειδί τη δράση Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το χρονικό διάστημα. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Πολλοί ζήτησαν ε, συμπληρωματική ερώτηση. Θα πρέπει να αποφασίσω ποιοι θα είναι οι δύο ομιλητέ οι οποίοι θα λάβουν το λόγο βάσει με, το, με τη σειρά που ζητήθηκαν ε, οι ερωτήσει και ποιο δεν έχει μιλήσει. Ο κύριο Ντέιβι και ο κύριο Όμπερμαϊερ. Ο κύριο Ντέιβι πρώτα, καταρχά. Ευχαριστώ. Ένα, μία από τι λίγε επιτυχίε τη Κοπενχάγη ήταν η συμφωνία για το μηχανισμό που θα διευκολύνει τις, ε, αναπτυσσόμενες, τις αναπτυγμένες χώρες να καταπολεμήσουν την καταστροφή των τροπικών δασών. Συμφωνείτε λοιπόν ότι μία από, τις, ε, από τους στόχους της Ισπανικής Προεδρίας θα είναι να δώσει ουσία στη συμφωνία αυτή και να διευκρινίσει από ευρωπαϊκής πλευράς τι είμαστε διτεθειμένοι να αφιερώσουμε για την αποτροπή της καταστροφής των τροπικών δασών. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για να πετύχουμε μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, εισήχθησε το σύστημα των πιστοποιητικών. Και αυτό θέλω να ρωτήσω. Πριν από λίγο καιρό ε, βγήκαν στο φως καταχρήσεις σε ό,τι αφορά την εμπορία των ρήπων. Θα εξεταστούν αυτές οι κατηγορίες και σε ποιο βαθμό προετοιμάζονται αλλαγές σχετικά με τις κατηγορίες αυτές. Ευχαριστώ, Υπουργός συμφωνώ με την πρώτη παρέμβαση. Νομίζω ότι ε, βρίσκεται στην κατεύθυνση και των δικών μα ε, συμπερασμάτων. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την καταστροφή των δασών στι αναπτυσσόμενε χώρε, γιατί αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη βελτίωση και τη ίδια τη ικανότητα αυτή ε, των αναπτυσσόμενων χωρών. Είναι λοιπόν προσφελώ η δράση αυτή. Και βεβαίω θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή των αυτόχθων πληθυσμών, των τοπικών πληθυσμών και η εγκατάσταση εθνικών συστημάτων ελέγχου των δασών. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι υπήρξε σημαντική πρόοδο στην Κοπενχάγη και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά το ζήτημα αυτό, αλλά και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, έχει παίξει ηγετικό ρόλο. Βρίσκεται ε, πρωτοπόρος. Οι επικρίσεις που μπορούσαν να, να αναφερθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Κοπενχάγη είναι ακριβώς ότι ε, ήταν πολύ πιο μπροστά από αυτό το οποίο επιτεύχθη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί πολύ περισσότερα και θέλει να εξεταστεί το θέμα σε πολύ περισσότερο βάθος. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με αυτά τα οποία είπατε. Ε, είναι θέμα το οποίο συνδέεται άμεσα με τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η συγκεκριμένη αυτή περίπτωση που αναφέρατε βεβαίως εντάσσεται σε αυτή την πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση των μέτρων καταπολέμησης της ε, κλιματική αλλαγή αποτελεί φυσικό και αναπόσπαστο τμήμα της όλης ε, διαδικασία, Πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου θα αποδυναμωθούν αυτές οι δράσεις επειδή ακριβώ γίνονται καταχρήσεις σε ορισμένα μέσα. Μα αυτό είναι ε, μέρος ε, της παθολογίας που να χαρακτηρίζει και το συγκεκριμένο αυτό μέτρο και άλλα. Ε, και θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτά. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ και τώρα θα περάσουμε στην επόμενη ερώτηση η οποία είναι... την έχει θέσει ο κύριος Aylward για τη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της νόσου του Αλτσχάιμερ. Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην νόσο του Αλτσχάιμερ και γενικώ στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Ο έλεγχος της νόσου αυτού θα πρέπει να είναι ένας κοινωνικός στόχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντικός πολιτικός στόχος. Ας μην ξεχνούμε ότι η εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ θα αυξηθεί εκθετικά ε, όσο γερνάμε και μετά τα 75 χρόνια διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Μάλιστα η Eurostat πιστεύει ότι ο αριθμός των ε, από την απτυνός Αλσχάιμερ θα διπλασιαστεί, ιδιαίτερα ως ένα 75 ετών. Η ερώτηση του κυρίου Άιλγουαρτ είναι δίπτυχη. Αφενός ε, μιλάει για μια πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού του Συμβουλίου για την καταπολέμηση των νευροεκφυλιστικών νόσων και αυτό σίγουρα έχει προβλεφθεί στο πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας που σας παρουσιάσαμε και ιδιαίτερα υπάρχει πρόβλεψη για την όσο του Αλτσχάιμερ. Και όπως ξέρετε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πρόταση που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, το Δεκέμβριο του 2009. Επίσης το Συμβούλιο έλαβε υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πιλωτική αυτή πρωτοβουλία του κοινού προγραμματισμού. Επίσης, σε ό,τι αφορά το συντονισμό της ε, ευρωπαϊκής δράσης, το Συμβούλιο πιστεύει ότι θα πρέπει να έχουμε πανευρωπαϊκή συνεργασία για την καταπολέμηση της νόσου Αλτσχάιμερ και συναφών ε, νόσων, γιατί θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μειώσουμε την επιβάρηση των ασθενών και των οικογενειών τους. Γιατί για κάθε άνθρωπο που υποφέρει από την νόσο αυτή υπολογίζεται ότι τρία μέλη της οικογένειας ε, ε, αναλαμβάνει το βάρος της φροντίδας του ασθενούς. Γι' αυτό και είναι απαραίτητη μια συνεργασία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην κοινή έκθεση για την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη που εθετήθηκε από το Συμβούλιο το 2008, τα κράτη-μέλη ανέλαβαν τη δέσμευση να αυξήσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να κάνουν έναν καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού κλάδου και τα κράτη-μέλη θεώρησαν ότι η παροχή υπηρεσιών ε, σε, στο σπίτι είναι προτιμότερη από ότι η παροχή υπηρεσιών στα νοσοκομεία. Βέβαια, οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είναι πρόκληση για πολλές χώρες μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς ε, χάραξε αυτούς τους αδρούς προσανατολισμούς για την αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ. Σας ευχαριστώ κύριος Άιλουαρτ. Ευχαριστώ Πρόεδρα και σας ευχαριστώ και σας Υπουργέ. Όπως είπατε, υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 ο αριθμός των ατόμων με άνοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πολλαπλασιαστεί και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει σωστή υποστήριξη για τους ε, για τα άτομα που τους, ε, για τους ε, θεραπευτές. Το ερώτημα λοιπόν που έχω να σας απευθύνω είναι πώς το Συμβούλιο θα υποστηρίξει συγκεκριμένα τα κράτη-μέλη προκειμένου η Άνια να καταστεί μια προτεραιότητα της ε, δημόσιας υγείας. Bien, eh, Η Ισπανική Προεδρία θέλει να προωθήσει τις εργασίες για μια κέρια σημασία οδηγία που θα αφορά τις προηγμένες θεραπείες και την παροχή φροντίδας σε χρόνιες νόσους ε, που δεν είναι μεταδοτικές. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και ταυτόχρονα θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας ε, και της ασφάλειας ε, της φροντίδας του ασθενού στην ομάδα εργασίας ε, υψηλού επίπεδου για τη δημόσια υγεία. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε και να δώσουμε τους προσανατολισμούς γιατί σε πολλές περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κατάλληλες αρμοδιότητες. Θα πρέπει να δώσουμε κάποιους ε, προσανατολισμούς και να προωθήσουμε τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών για να υπάρξει μια κοινή αντιμετώπιση αυτών των νευροεκφυλιστικών ασθενειών και κυρίως ε, της νόσου Αλτσχάιμερ. Επίσης, θα πρέπει και έμεσα να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη, γιατί τα κράτη-μέλη είναι αυτά που φέρουν την ευθύνη της παροχής πιο άμεσης ενίσχυσης προς τις οικογένειες ή προς μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Βέβαια, σε ένα ε, δημόσιο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Υγείας ε, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε κάποια ταμεία και κονδύλια και έτσι έστω και έμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει τους ε, πάσχοντες ή τις οικογένειές τους γιατί οι πάσχοντε πραγματικά είναι εξαρτημένοι από τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα όταν πάσχουν από Αλσχάιμερ ή άλλες νευροεκφυλιστικές νόσους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δύο συμπληρωματικέ ερωτήσεις από τον κύριο Χίγγινς και την κυρία Τικάου. Πρώτο ο κύριος Χίγγινς. Ευχαριστώ πρόεδρε και να ευχαριστήσω και το Συμβούλιο για την απάντηση. Να ρωτήσω το εξής. Ποια η στάση σας σε ό,τι αφορά την ε, λήψη τροφής παραντερικά των ασθενών. Είναι σημαντικό να υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες. Αυτό, αυτή η διαδικασία δίνει ε, παρκή τροφή στον ασθενή σε περίπτωση που αρνούνται την πρόσληψη τροφής λόγω άνοιας. Σκοπεύετε να θέσετε σχετικά πρότυπα. Ευχαριστώ, κυρία Τικάου. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες επηρεάζουν δυστυχώς πολλούς ανθρώπους και σε ορισμένες χώρες δεν υπάρχουν αρκετές ε, δυνατότητες ε, έγκαιρης διάγνωσης ή παροχής φροντίδας ε, και θεραπείας ε, στους πάσχοντες. Θα θέλετε να δημιουργηθούν κάποια ευρωπαϊκά κέντρα θεραπείας που να μπορούν να παράσχουν φροντίδα σε πολλούς ασθενείς και επίσης να προωθήσουμε και ερευνητικά κέντρα που θα αναζητούν φάρμακα για τις νευροεκφυλιστικές νόσους. Ο κύριος Υπουργός. Κύριε Πρόεδρε. Στις δύο συμπληρωματικές σας ερωτήσεις θα πρέπει να αναζητήσουμε κάποια επιστημονική απάντηση. Και από αυτή την άποψη υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ομάδες και πρωτοβουλίες που είναι πιο κατάλληλες και αρμόδιες για να δώσουν απαντήσεις στα ειδικευμένα σας ερωτήματα. Για παράδειγμα, υπάρχει το πιλωτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση των νευροεκφυλιστικών νόσων και ιδιαίτερα της νόσου Αλσχάιμερ. Για το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για σύσταση προς το Συμβούλιο που έχει ήδη δρομολογηθεί και όπως ξέρετε και σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει και μια ομάδα υψηλού επίπεδου για τον κοινό προγραμματισμό για την καταπολέμηση αυτών των ασθενειών, που είναι χρόνιες, επαναλαμβάνω, και μη μεταδοτικές. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εκ του την εφαρμογή αυτής της πειραματικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν και να προσδιοριστούν κάποια θέματα και να διευκολυνθεί η λήψη πιο συγκεκριμένων αποφάσεων, όπως αυτές που ζητήσατε εσείς με τις συμπληρωματικές σας ερωτήσεις. Και νομίζω ότι σε αυτά τα φόρα θα πρέπει να εξεταστούν όλα αυτά τα θέματα. Η ομάδα υψηλού επίπεδου αυτή τη στιγμή ασχολείται με το στρατηγικό πρόγραμμα για την έρευνα Συμμετέχουν εκεί 24 χώρες και τώρα προσδιορίζονται οι, οι διαχειριστικές διαρθρώσεις και το πρόγραμμα εργασιών. Μάλιστα θα υποβάλει αυτή η ομάδα υψηλού έκθεση προς την Ισπανική Προεδρία και μετά την έκθεση αυτή θα υποβληθούν πιο συγκεκριμένες προτάσεις για αυτές τις λύσεις. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ομάδα υψηλού και οι αντίστοιχες δομές για να επεξεργαστούν όλα αυτά τα θέματα και να προλιάνουν το έδαφος για τη λήψη αποφάσεων. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ, Υπουργέ. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Χίγκινς δεν θα έχει ικανοποιηθεί με την απάντηση αυτή, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο το θέμα αυτό και προφανώς ε, αξίζει να ρωτηθεί από μόνο του σε κάποια φάση. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο, στην επόμενη ερώτηση του κυρίου Ντεζίρ αναφορικά με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός. Πρέπει να αναφερθώ στη διάσκεψη για την ε, κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων που έγινε στη Στοχόλμη στις 10 και 11 Νοεμβρίου του 2009. Ε, η Σουηδική Προεδρία, η οποία διοργάνωσε αυτή τη διάσκεψη και η τότε επόμενη Προεδρία, σήμερα ε, τρέχουσα Προεδρία, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όσον αφορά το ζήτημα αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει να, να δώσει το παράδειγμα στο συγκεκριμένο αυτό θέμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο θέτει και με την ερώτηση του κ. Δεζίρ η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων ε, όταν μιλάμε για τη δημιουργία αγορών, καταπολέμηση διαφθοράς, ε, υποστήριξη του περιβάλλοντος, προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην, ε, στον, τόπο, χώρο της εργασίας, μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είμαστε η πιο σημαντική οικονομία στον κόσμο. συμβάλλουμε περισσότερο από του υπόλοιπου στη συνεργασία για την ανάπτυξη. Έχουμε πολλέ πολυεθνικέ εταιρείε. Ε, άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι το κατάλληλο επίπεδο στο οποίο πραγματικά θα πρέπει να αναλυφθεί και η ευθύνη για την αντιμετώπιση του ζητήματο. Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων έχει τρει συνιστώσει. Protect, respect, remedy. Προστασία, σεβασμός, ε, επανόρθωση. Προστασία σημαίνει νομοθεσία, ε, για παράδειγμα στο θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως στον αφορά το ζήτημα αυτό από τις επιχειρήσεις. Επίσης υπάρχει η εταιρική ευθύνη για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευθύνη όλων των εμπλεκομένων μερών για να υπάρξει η δυνατότητα επανόρθωσης επαρκούς. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε άλλο ένα μέσο στη διάθεσή μας που είναι η Χάρτα των ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, των ε, Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα μέσο το οποίο είναι νομικά δεσμευτικό και για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει, θεσπίζεται μάλλον αυτή η προστασία για τα θέματα αυτά στα οποία αναφέρεται και ε, η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να εξακολουθήσει ο διάλογο με τα κρατημέλη, με την κοινωνία των πολιτών, με τα συνδικάτα, με τι επιχειρήσει και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, έτσι ώστε να ε, ολοκληρωθεί αυτή η τριλογία ε, του Protect, Respect and Remedy. Η Ισπανική Προεδρία θα εξακολουθήσει να προωθεί το θέμα αυτό. Μάλιστα, στην Πάλμα de Μαγιόρκα στι 25 και 26 Μαρτίου θα διοργανώσει διάσκεψη που θα εξετάσει το ζήτημα τη θεσμοθέτηση τη κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων από τη σκοπιά ε, των σχέσεων με τον, ε, ε, με τον εταιρικό διάλογο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν τα κατάλληλα μέσα έτσι ώστε να προωθήσουμε και να εφαρμόσουμε αυτέ τι δραστηριότητε και μάλιστα και σε σχέση με κάτι το οποίο αναφέρθηκε σήμερα το πρωί κατά την παρουσίαση του προγράμματος της Ισπανική Προεδρία Η στρατηγική για το 2020. Και εδώ εντάσσεται άμεσα και το θέμα του στόχου της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε τον Υπουργό, κύριε Στυζήρ. Σας ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε Υπουργέ για την ε, ε, απάντησή σα, Σας συγχαίρω για αυτή τη διάσκεψη που θα γίνει το Μάρτιο στην Παλματέ Μαγιόρκα που θα αποτελέσει τη συνέχεια της διάσκεψης στο Κόλμη. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πολυεθνικές. Το είπατε. Πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο η Ευρώπη στο θέμα αυτό. Αλλά... Ε, τι γίνεται και με τη συμπεριφορά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εκτό ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση Μιλούμε για τι θηγατρικέ ε, των ε, εταιριών αυτών που έχουν διαφορετικό νομικό πρόσωπο. Σκέφτεστε κάποιο νομικό μέσο όπου η μητρική επιχείρηση θα αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμπεριφορά των θηγατρικών και των υποκαταστημάτων στα υπόλοιπα σημεία τη γη, όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων κτλ. Διαφορετικά η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων που θέλει να προωθήσει η Ευρώπη θα μα οδηγήσει οδηγεί σε μια κατάσταση όπου θα, θα ξεφεύγουν οι επιχειρήσει από τον έλεγχο λόγω τη δημιουργία ε, θηγατρικών ε, σε άλλα σημεία τη γη εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε, Υπουργό. Ναι, νομίζω ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να, να, να προωθήσει ε, τις βέλτιστες πρακτικές. Και Μάλιστα, για αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρξουν οι απαραίτητε νομοθετικέ προτάσει για να βελτιώσει την κατάσταση. Όσον αφορά το θέμα τη κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, μην ξεχνάμε ότι έχει μία συνιστόσα που είναι νομικά δεσμευτική, α την πούμε έτσι, και που έχει να κάνει με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά έχει και ένα, μία συνιστόσα εθελοντική φύση, μέσα δηλαδή από εθελοντικέ πρακτικέ. Γι' αυτό αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να δημιουργηθούν τα κατάλληλα φόρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέραν των υφιστάμενων, έτσι ώστε να εξεταστούν αυτέ οι πτυχέ. Ήδη έχουν ξεκινήσει ορισμένε πρωτοβουλίε προ την κατεύθυνση αυτή. Και μάλιστα, να σα αναφέρω το εξή. Για παράδειγμα, η ομάδα υψηλού επίπεδου των κρατών μελών συνεδριάζει κάθε έξι μήνε για να υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών στο ζήτημα αυτό της ε, κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Και επιπλέον πιστεύω ότι στα πλαίσια αυτά, ε, στα σημερινά πλαίσια της οικονομικής κρίσης, ε, το θέμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Μην ξεχνάμε ότι το 2010 είναι το έτος καταπολέμησης της στόχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση της κατεύθυνσης που θα ακολουθήσουμε. Και κάτι άλλο, μην το ξεχνάμε, με βάση αυτή την πρωτοπόρα εκδήλωση θα πρέπει να δημιουργήσουμε και άλλα φόρα όπως σας είπα. Εκεί όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι οι stakeholders όπως λέμε, θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα διάλογο, διάλογο που θα, από τον οποίο θα πρέπει να υπάρξουν τα μεταγενέστερα μέτρα. Πάντω χρειάζεται αυτή η φάση διαλόγου που είναι απολύτω ουσιαστική ε, σημασία ε, για κάτι στο οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Και τώρα έχουν ζητήσει πάλι τη συνάδελφοι το λόγο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κόζα και στον κύριο Μάρτιν. Γιατί είναι η πρώτη φορά που ζητούν το λόγο. Ο κύριος Κόζα, λοιπόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόζα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Υπουργό και μου άρεσε κάτι από αυτά που είπε. Όλοι ξέρουμε ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γυράσκει και ότι οι επιχειρήσεις φέρουν ευθύνη για τα άτομα εκείνα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την, την των ατόμων αυτών στην κοινωνία, γιατί είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη η συμβολή τους. Danke. Ο κ. Μάρτιν, ευχαριστώ. Το ερώτημα... Τα ερωτήματα που θίξατε μας απασχολούν εδώ και πάρα πολύ καιρό και πολλά από αυτά που ακούσαμε θα μπορούσαμε να τα έχουμε ακούσει και πριν από 10-15 χρόνια. Συγκεκριμένες ερωτήσεις λοιπόν, συμφωνείτε μαζί μου. Για την προαγωγή της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων χρειάζονται κίνητρα αλλά και κυρώσεις. Επίσης, μπορείτε να φανταστείτε ένα σύστημα naming and shaming δηλαδή που θα κατανομάζουμε τους υπεύθυνου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί βλέπουμε πόσο συχνά υπάρχουν επιγραφές, ετικέτες ε, σήμερα. Θεωρείτε ότι αυτό συνάδει με την ε, κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Έχουμε συνηθίσει τόσες πολλές ετικέτες. Γιατί να μην γίνεται αυτό και στον κοινωνικό τομέα. Ευχαριστώ για να απαντήσει ο Υπουργός. Συμφωνώ με την πρώτη παρέμβαση, με την έννοια ότι πράγματι στο βάθος και πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο διάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα, με τα με την κοινωνία των πολιτών, με τα συνδικάτα και με όλους τους εμπλεκόμενους. Η συμμετοχή λοιπόν όλων αυτών που αναφέρατε και εσείς είναι απολύτως ουσιαστική σημασία. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια ε, κρίσιμη στιγμή όπου πρέπει να σκεφτούμε το ζήτημα αυτό και πρέπει να σκεφτούμε και αυτό το οποίο είπατε κι εσείς. Βεβαίως. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι στα πλαίσια μιας συνολικής προσέγγισης ε, του ζητήματος ίσως για πρώτη φορά ή σχεδόν για πρώτη φορά νομίζω ότι πρέπει να επιδείξουμε μεγάλη αποφασιστικότητα. Και υπάρχει μέσω αυτή τη ομάδα υψηλού επίπεδου, αλλά και μέσω αυτή τη διάσκεψη που θα γίνει το Μάρτιο. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να ε, σταθούμε και να προβληματιστούμε σε βάθος και, ο και αυτό αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να πετύχουμε τους στόχους μας. Μερικές φορές ε, η βέλτιστη οδός είναι τα κίνητρα, άλλες φορές οι κυρώσεις. Δεν είναι πάντα όμω οι κυρώσει ε, ο βέλτιστο δρόμο. Θα πρέπει να μελετηθούν όλα τα στοιχεία. Και αυτό το οποίο απαιτείται είναι ολοκληρωμένη θεώρηση και εξέταση και μία σειρά μέτρων που δεν είναι σπασμωδικά ή ε, ε εξατομικευμένα, αλλά επιτέλους να υπάρξει μία ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνολικού ζητήματος. Γιατί έχουμε μία θαυμάσια ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ. Υπουργέ, και τώρα περνάμε στην επόμενη ερώτηση, στην ερώτηση του κυρίου Μάρτιν αναφορικά με την χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Μάρτιν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μία σοβαρότατη χρηματοπιστωτική κρίση. Αλλά προσπαθεί να επιβάλλει μία πραγματική ρυθμίση χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα αυτό το κάνει μέσω δύο διαστάσεων που περιλαμβάνονται στις έξι οδηγίες χρηματοπιστωτικής εποπτείας και που υπέβαλε πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση διαβούλευσης μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Ισπανική Προεδρία είναι υπέρ της επίτευξης συμφωνίας επί των οδηγιών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και σημαντικός διαμεσολαβητής εδώ και συνομιλητή μας θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα για το για τη μακροπροφυλακτική εποπτεία είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την αποτροπή του συστημικού κινδύνου, γιατί χάρη στα μέτρα αυτά προσπαθούμε να αποτρέψουμε σημαντικές κρίσεις, να μειώσουμε τις διαταραχές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να αποκαταστήσουμε μια σταθερότητα. Και έχουμε και τη μικροπροφυλακτική εποπτεία είναι αυτή στην οποία αναφέρεται στην ερώτηση του κυρίου ε, Hans Peter Martin. Είναι οι τρεις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τράπεζες, τις, ασφαλεί, ασφάλειες και τις α, ε, ε, χρηματαγορές ή τις αγορές αξιογράφων. Χάρη στις διατάξεις αυτές θα επισέλθουμε στα βαθιά νερά της εποπτείας μέσω της μείωσης των διαταραχών και στα μεμονωμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φορείς. Και έτσι θα προστατεύσουμε τους πελάτες αυτών των χρηματοπιστωτικών φορέων. Το Συμβούλιο, όπως σας είπα, έχει εγκρίνει οριστικά την κοινή του θέση. Πρώτα στο περσινό Συμβούλιο που έγινε τον Οκτώβριο. Εκεί έγινε δεκτή η συμφωνία, η πολιτική συμφωνία επί της αρχής για την μακροχρηματοπιστωτική εποπτεία και το Δεκέμβριο εγκρίθηκε η μικροχρηματοπιστωτική εποπτεία με το σύνολο του νομοθετικού πακέτου. Επαναλαμβάνω ότι οι οδηγίε αυτέ εμπίπτουν στη διαδικασία τη συναπόφαση. Γι' αυτό και θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Πάντω, οι τρει επιτροπέ θέλουμε να λειτουργήσουν το συντομότερο δυνατόν και μακάρι οι οδηγίε να εγκριθούν ήδη κατά το εξάμεινο τη Ισπανική Προεδρία. Πάντω, θέλουμε οι επιτροπέ αυτέ στα τέλη τουλάχιστον το 2010 να έχουν μπει στι ράγες και να είναι ήδη λειτουργικέ. Αυτό είναι ο στόχο του Συμβουλίου. Και προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διεκπαιρεώσουμε αυτό το σημαντικό ποιοτικό άλμα που θα είναι και ιστορική σημασίας. Ανταποκρίνεται άλλωστε ε, σε προηγούμενους προσανατολισμού του G20, γιατί και οι Ηνωμένε Πολιτείε εφαρμόζουν αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση και αυτή είναι η σημαντική μας πρόκληση για να αποτρέψουμε στο μέλλον μια παρόμοια κρίση με τη σημερινή που εκπορεύθηκε από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, την έλλειψη ρύθμισης που το χαρακτήριζε και την ανευθυνότητα, όπως είπε και κάποιος προλαλή σας, κάποιων ε, ηγετικών στελεχών αυτού του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Αναφερθήκατε στον ε, μακροοικονομικό τομέα. Θα γνωρίζετε βέβαια ότι υπάρχουν έντονες κριτικές σε ό,τι αφορά το σχετικό συμβούλιο και το μέγεθός του. Θεωρείτε, όπως πολλοί άλλοι, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορέσει να εργαστεί τόσο αποτελεσματικά όσο θα έπρεπε και κατά δεύτερον τίθεται και θέμα ανεξαρτησίας ε, του Συμβουλίου αυτού της Επιτροπής αυτής. Θεωρείτε ότι η Ισπανική Προεδρία θα κάνει ένα βήμα παραπέρα για να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της Επιτροπής αυτής και σε ό,τι αφορά να, το θέμα του, της σύνθεσης, του μεγέθους της Επιτροπής να τη βελτιώσει για να είναι πιο αποτελεσματικό το έργο της. Minister. Ευχαριστώ, Υπουργός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση και υπήρξε συμφωνία, η συνένεση στο Συμβούλιο. Μια πολιτική συμφωνία που δεν ήταν καθόλου εύκολη, γιατί χρειάστηκε να επιμείνουν και η Σουηδική Προεδρία και η Επιτροπή στο ΕΚΟΦΗΝ για την επίτευξη αυτής της συνένεσης. Τώρα υπάρχει αυτή η απόφαση, η κοινή θέση του Συμβουλίου και φτάνει το θέμα στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο θα συζητήσει τη συμφωνία αυτή και ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί συμφωνία. Γιατί υπάρχει μια συνένεση στο Συμβούλιο, θα δούμε πώς ε, θα επιτύχουμε και συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το θέμα αυτό είναι αντικείμενο συζήτηση όπω και άλλα. Πάντω είμαι βέβαιο ότι θα καταλήξουμε στη συμφωνία, γιατί είναι απολύτω απαραίτητη η συμφωνία μεταξύ των δύο νομοθετικών βραχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Έχουμε και πάλι πολλές συμπληρωματικές ερωτήσεις. Πάντα ακολουθώ το κριτήριο του ποιος δεν έχει μιλήσει και ποιος ζητάει πρώτο το λόγο. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Κέλλη και στον κύριο Χουντή. Ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μέρος ε, των προτινόμενων μέτρων εποπτείας, χρηματοοικονομικής εποπτείας. Η Ισπανική Προεδρία θα εξετάσει την ε, θέσπιση ενότατου ορίου των αμοιβών των ε, υψηλών στελεχών που οδήγησε εν μέρει στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Κύριε Σχουντής. Ναι. Κύριε Υπουργέ, θέλω να συνδέσω το θέμα της χρηματοπιστωτικής εποπτείας της ευρωπαϊκής ένωσης με την κερδοσκοπική δράση που αναπτύσσουν εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων που μάλιστα εδρεύουν στην ευρωπαϊκή ένωση στο city του λονδίνου. δημοσιεύματα λένε ότι ε, ε, διαχειριστές τέτοιων εταιριών ποντάρουν πτωτικά στο ευρώ στα δημόσια ομόλογα της ελλάδας και αλλού στο χρέος και στο έλλειμμα με συνέπεια να επιδεινώνεται ο δανεισμός είσαστε σε θέση λοιπόν να μου πείτε τι συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να ληφθούν ούτω ώστε να προστατευτούν οι οικονομίε των χωρών μελών της ευρωπαϊκής Ένωση από τι κερδοσκοπικέ επιθέσεις των εταιριών αμοιβαίων κεφαλαίου υψηλού ρίσκου που μάλιστα εδρεύουν στην ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ. Thank you very much, Minister. Ο Υπουργός έχει λόγο. Bueno, yo creo que sí que... Φυσικά. Και είναι δυνατόν να συζητήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φορείς. Και ξεκινάει μια συζήτηση που περιστρέφεται γύρω από τα διάφορα συστήματα χρηματοπιστωτικής εποπτείας και εδώ είναι η κατάλληλη ευκαιρία και το κατάλληλο φόρουμ για να επεξεργαστούμε αυτό το θέμα και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες ε, οδηγίες που θα καλύπτουν όλα αυτά τα στοιχεία που επισημάνατε κύριε Κέλλη. Και η πρόταση που μας έκανε ο δεύτερος ομιλητής εντάσσεται σε αυτές τις οδηγίες που θα εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την οδηγία για την ε, ρυθμίση των hedge funds, για παράδειγμα, που και αυτά θα πρέπει να καλυφθούν από τις ανάγκες εποπτείας. Ή σε κάτι που ανέφερε το πρωί ο Προεδρεύων της Ένωσης, το θέμα της ε, κατάργησης των φορολογικών παραδείσων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι ιδέες που προτάθηκαν και μπορεί να είναι αντικείμενο της συζήτησης που θα γίνει τους επόμενους μήνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να καταλήξουμε σε μια μεταρρύθμιση που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη χαρακτήρισε ως πλήρη και πραγματική μεταρρύθμιση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μια ευρυθή και διεξοδική μεταρρύθμιση στην οποία θα αναλυθούν όλες αυτές οι προσεγγίσεις και όλες αυτές οι λύσεις. Σας ευχαριστώ, Υπουργέ, και τώρα περνάμε στην επόμενη ερώτηση του κυρίου, της κυρίας Κράτσα που αφορά την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, τη δημοσιονομική κατάσταση στην Ελλάδα και το ρόλο της Ευρωζώνης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, υπάρχει σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων. Οι οικονομικές πολιτικές ε, των κρατών μελών είναι βεβαίως κάτι που ενδιαφέρει από κοινού την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ταυτόχρονα οι εθνικοί προπολογισμοί είναι εθνική αρμοδιότητα. Και ακριβώς γι' αυτό, δεδομένου βεβαίως ότι υπάρχει στις 16 χώρες ένα κοινό νόμισμα, και ταυτόχρονα προβλέπεται διεύρυνση γιατί η ιδέα της νομισματικής ένωσης είναι κάτι που ε, συμπεριλαμβάνεται στη θήκη του Μάστριχτ ως ε, ε, στόχος όσο το δυνατόν γενικότερος καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες από τα κράτη σε σχέση με τους προπολογισμού τους, διότι η δράση τους επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας και του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος. Γι' αυτό πρέπει να αποφεύγονται τα υπερβολικά δημόσια ελλείμματα. Και αυτό είναι ουσιώδης σημασία για τη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και βεβαίω πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ε, με βάση όλα αυτά ε, λειτουργήσε η Νομισματική Ένωση. Εξού και το Σύμφωνο της σταθερότητα, και εξού και το γεγονός ότι σήμερα στη συνθήκη λειτουργίας ε, ε της Ευρωπαϊκής Ένωσης 123, στο άρθρο 23, ε, αναφέρονται, ε, αναφέρεται η δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, και το θέμα των δανείων. Επίσης, αναφέρεται στην Ένωση, στην συνθήκη, ότι ούτε τα κράτη-μέλη, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπόλογοι για τη δράση του κάθε κράτους μέλους. Γι' αυτό με δύο λόγια. Ε, κάθε κράτο μέλο ε, πρέπει να αντιμετωπίσει μόνο του τι υποχρεώσει του στον τομέα του χρέου και ε, αυτό ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Εξακολουθεί λοιπόν να πιστεύει το Συμβούλιο ότι και η Ελλάδα αλλά και τα υπόλοιπα θα λάβουν τι απαραίτητε ε, και τι σωστέ αποφάσει για να αποφύγουν ε, αυτή την έλλειψη ισορροπία και να υπάρξει παγίωση των ε, οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πλαισίων σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η διαδικασία του υπερβολικού δημοσιονομικού ελέγχου, του δημοσιονομικού ελλείμματο, προβλέπει εποπτεία σε περίπτωση που δικαιολογείται κάτι τέτοιο. τώρα, το Συμβούλιο θα συζητήσει την περίπτωση τη Ελλάδα, πιστεύω, το Φεβρουάριο. Και είναι πιθανό τότε Βεβαίω, έχει δικαίωμα πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, και ε, είναι πιθανό να υπάρξουν υποδείξει και συστάσει και να εξεταστούν ε, στρατηγικέ. Γιατί με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της και την εμπλοκή της σε τέτοιες περιστάσεις ε, δυσκολίας, όπως αυτές που αντιμετωπίζουν διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ... Περιμένω Ευχαριστώ ε, κύριε Προεδρεύοντα για την απάντησή σας. Υπενθυμίσατε τις, τα άρθρα τη της συνθήκης που αντιστοιχούν στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος γνωρίζει το κοινοβούλιο τα άρθρα αυτά αλλά έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσατε να με, πληροφορήσετε τι εννοεί ο κύριος Θαπατέρο όταν λέει για αλληλεγγύη στην Ευρωζώνη, για αλληλεγγύη σε χώρες με ιδιαίτερα δημοσιονομικά προβλήματα. Μήπως υπάρχει το ενδεχόμενο της συζήτησης ενός καλύτερου δημοσιονομικού συντονισμού μεταξύ κέντρου και περιφέρειας όσον αφορά τις επιδόσεις μήπως καλύτερου φορολογικού συντονισμού για να αποφευθεί το dumping το φορολογικό το κοινωνικό που ήδη επιβαρύνει την ευρωπαϊκή ένωση και έχει ε, συνέπειες ιδιαίτερες σε κάποιες χώρες. Ε, κάτι παραπάνω μπορείτε να μου πείτε από αυτό που αναφερθήκατε και προφανώς εννοεί ο κύριος θαπατέρο αλληλεγγύη. ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο Υπουργό. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ε, περιοχή ε, στον κόσμο, αν θέλετε, όπου η αλληλεγγύη ασκείται με πολύ ορατό τρόπο. Για παράδειγμα, όσον αφορά την Ελλάδα ε, ή όσον αφορά τη χώρα μου, την Ισπανία. Πρέπει να σας πω ότι εμείς ε, είδαμε τη μεγάλη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, μέσα από τα ευρωπαϊκά ταμεία, τα διευθυντικά ταμεία. Όλα αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία της πολιτικής της αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα στοιχεία αυτά δεν, ε, ε, αυτό ε, είναι κάτι το οποίο δεν εμφανίζεται αλλού σε άλλη γωνιά της γης. Και αυτό οδήγησε σημαντική πρόοδο σε, σε πολλές χώρες και αυτό ωφελεί ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άνοιγμα των αγορών, για παράδειγμα, καθώς επίσης μεταφορά συγκεκριμένων κονδυλίων και τον εξυγχρονισμό μια συγκεκριμένη περιοχή, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο, εξαιρετικό παράδειγμα αλληλεγγύη. κονδύλια, τα οποία βεβαίω πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωστά και γι' αυτό προβλέπονται και έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα το οποίο απολύτω λογικό και φυσικό. Άρα αλληλεγγύη υπάρχει. Και μία μορφή αλληλεγγύη επίση είναι αυτό το οποίο αναφέρεται και μέσα στη συνθήκη. Ναι, μια και αναφερθήκαμε στη συνθήκη. Στη συνθήκη αναφέρεται η υποχρέωση των κρατών μελών να συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές, τις κοινωνικές πολιτικές και τι πολιτικέ στον τομέα τη απασχόληση το άρθρο 5 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αναφέρει με σαφήνεια και εκεί επίσης εκφράζεται η αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκή Ένωση, στον κοινό προβληματισμό και στην κοινή υιοθέτηση στόχων εν ώψη μιας οικονομικής πολιτικής που θα πρέπει να είναι συντονισμένη. Πολλά από τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν διάφορες χώρες της Ευρώπης ως συνέπεια της κρίσης δεν θα είχαν υπάρξει ή τουλάχιστον δεν θα ήταν τόσο έντονα αν υπήρχε οικονομική ένωση πολύ νωρίτερα γιατί η Οικονομική ε, ε, Ένωση ε, σταμάτησε και δεν υπήρξε αυτή η συνέργεια συντονισμού των οικονομικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε σε τελευταία ανάλυση. Και αυτό προτείνεται μέσα από τη συνθήκη η στρατηγική της Ευρώπης για το 2020, οι στόχοι που θα πρέπει να είναι κοινοί μας στόχοι και που αφορούν τις επενδύσεις, την εκπαίδευση, στην παιδεία, στην εξειδίκευση των εργαζομένων, στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και αυτά είναι στοιχεία κοινά, τα οποία εκφράζουν την αλληλεγγύη όλων μας και με τον τρόπο αυτό εκφράζεται ιδιαίτερα η αλληλεγγύη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ενωμένη, όλο και περισσότερο ενωμένη. Και βεβαίως αυτό δεν εμποδίζει η συνθήκη με αρκετά ε, ξεκάθαρο τρόπο να απαιτεί ανάληψη ευθύνης από εκ μέρους των κρατών μελών όσον αφορά το επίπεδο του χρέους τους ή ε, τι ε, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι αρμοδιότητα κάθε κράτο μέλους. Αλλά όλα αυτά μέσα στα πλαίσια μια αγορά κοινωνικών πολιτικών, διευθυντικών πολιτικών, περιφερειακών πολιτικών και στο μέλλον ελπίζω συντονισμού των οικονομικών, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών στον τομέα τη απασχόλησης. Γιατί αυτό είναι ένα περιβάλλον, ένα πλαίσιο ελληνική. Είναι ο πιο σωστό τρόπο για να ε, εφαρμόσουμε την πολιτική αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε e, Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Γιατί είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι η κατάσταση στην Ελλάδα είναι δεινή και ότι θα απασχολήσει την ε, Επιτροπή το Φεβρουάριο. Σίγουρα υπάρχει σοβαρή κρίση εντός της Ελλάδας, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι δεν ξέρουμε πώς θα λυθεί. Το θέμα είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να γίνει μία συζήτηση ουσιαστική και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σημαντικό θεσμικό όργανο και θα πρέπει ίσως να δραστηριοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί περισσότερο και για την κατάσταση στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Bueno, eh, Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι κάθε όργανο και κάθε θεσμός έχει τη, ε, τους δικούς του τομείς εργασίας και αυτό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά ε, της δομής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης στην Ευρώπη. Και αυτό άλλωστε της προσδίδει την αξιοπιστία, προσδίδει την αξιοπιστία στην Ένωση. Είναι σαφές ότι το Συμβούλιο θα ασχοληθεί με την περίπτωση της Ελλάδας γιατί πρόκειται για ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εταίρο μας, και ε, αφορά όλους αυτή η κατάσταση. Προφανώς ε, αυτό το οποίο συμβαίνει σε μια άλλη ε, χώρα μέλος μας αφορά. Ε, γιατί εδώ μιλάμε για μια ε, εσωτερική αγορά και για 16 ένα κοινό νόμισμα για 16 χώρες. Στα πλαίσια λοιπόν και στα όρια που θέτει η συνθήκη θα συζητηθεί το ζήτημα αυτό και ταυτόχρονα θα συζητηθεί η δημοσιονομική στρατηγική που θα θεωρηθεί ε, η σωστή υπό τις παρούσες συνθήκες και που θα υποδειχθεί εμπροκειμένω στην Ελλάδα. Και βεβαίως η Ελλάδα θα ωφεληθεί από όλες αυτές τις υποδείξεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, έχει τις συγκεκριμένε αρμοδιότητες που περιγράφονται στη συνθήκη όσον αφορά την νομισματική σταθερότητα και όσον αφορά την σταθερότητα των τιμών μέσα σε ε, όρους ανεξαρτησίας. Η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί ουσιαστική αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η αρχή επιτρέπει ε, το οικονομικό και νομισματικό μας σύστημα να χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη αξιοπιστία και το νόμισμά μας, το ευρώ. Αυτό το κριτήριο λοιπόν τη αμεροληψία και τη ανεξαρτησία πρέπει να είναι σεβαστό και να τηρείται γιατί αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό του οικοδομήματο νομισματική και οικονομική ένωση που αποφασίσαμε πριν λίγα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank Σας ευχαριστώ Υπουργέ, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας αυτή την πρώτη, ε, στο πρώτο γύρο ερωτήσεων της Προεδρίας. Ε, Ελήψη χρόνου, οι υπόλοιπε ερωτήσεις θα απαντηθούν εγγράφως και ε, διακόπτονται η συνεδρίαση μέχρι τις 9 το βράδυ.